στον οποίο παραλάβαμε την εμπιστοσύνη μας, ε, για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, ενωμένοι και με διαφάνεια. Αυτά είναι σημαντικά κλειδιά, όπως έχουμε ξαναπεί, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να στεφθούν με επιτυχία. Ε, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθημερινά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Φυσικά, ε, γνώμονάς μας θα είναι πάντα ίσοι κανόνες παιχνιδιού και για τα επόμενα στάδια της διαπραγμάτευσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προθεσμίες που πιέζουν και διαδικασίες που πρέπει να μας απασχολήσουν ε, κατά το θέρος, αν ζητηθούν παρατάσεις. Πάντω σήμερα δεν έχουμε την πρόθεση να προεξοφλήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ας αρχίσουμε από την αρχή, δηλαδή το συντομότερο ε, να ε, κατοχυρωθεί το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να αποφανθεί για την αποχώρηση και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα υπηρετήσουμε καλύτερα το ευρωπαϊκό συμφέρον πάντα σε πάρα πολλή συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία σε θέματα οικονομικά, εμπορικά αλλά και ασφάλειας και άμυνας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ασχοληθούμε με το ζήτημα της διάσκεψης αυτής για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, αναφέρθηκαν πολύ προηγουμένως ε, στη συζήτηση για την επέτειο της Ενδείξης Λισαβόνας. Αυτό το θέμα το Συμβούλιο το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Κατανοούμε τις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών. Θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο. Να μην θεωρήσουμε ότι στα διάφορα κράτη ή στην Ευρώπη αυτό που μας ενδιαφέρει να ψηφίζουμε κάθε 4-5 χρόνια και μετά οι πολίτες να είναι παθητικοί θεατές των αποφάσεων που τους αφορούν. Κατανοούμε αυτό το μέλημα των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων προφανώς και η επιθυμία μας είναι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, να είμαστε ε, καλόπιστοι, ε, αφοσιωμένοι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά λέμε ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρακαλώ κατανοήστε το αυτό, έχει σημασία να κρατήσει τη δυνατότητα δράσης του βράχη πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα για τα στρατηγικά ζητήματα θέλει το Συμβούλιο να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει να προωθεί αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Είχαμε πει στην ευκαιρία να συζητήσουμε τις διεθνείς σχέσεις με ιδιαίτερη εστίαση στο θέμα της Τουρκίας και την εκεί κατάσταση. Δεν έγινε εκτεκταμένη συζήτηση για την Τουρκία. Του χρόνου θα έχουμε πιο στρατηγική συζήτηση για τα γενικά γεωπολιτικά ζητήματα. Πάντως διατρανώσαμε και πάλι απερίφραστα ε, την απόλυτη αλληλεγγύη μας με την Ελλάδα και την Κύπρο, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων που γνωρίζετε. Τέλος, δύο λόγια για την Ατζέντα 2020, αυτό το θεματολόγιο. Θέλησα να παρουσιάσω μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια μέθοδο εργασίας και μια στρατηγική ατζέντα για το 2020 για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε του χρόνου. Θα πρέπει να αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτά είναι το κλίμα, όπως έχετε καταλάβει, θα παραμείνει κυρίαρχο ε, στο πολιτικό θεματολόγιο για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επίσης, το ψηφιακό θεματολόγιο θα είναι σημαντικό θέμα. Την ε, Άνοιξη θα έχουμε μια σύνοδο κορυφής ε, κάποια χρόνια μετά το Ταλίν και της ευρεία εφαρμογής του, θα πρέπει τώρα να ασχοληθούμε ξανά με αυτό το θέμα. Έχουμε μεγάλη φιλοδοξία για τα big data, για την ε, τεχνολογία 5G, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να είμαστε και εκεί πρωταγωνιστές. Το θέμα το μεταναστευτικό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επανέλθει και το 2020 επιτάπητος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και φυσικά όλα τα ζητήματα ασφαλείας και άμυνας είναι εκ των όν ουκ Γιατί συνδέονται με την δυνατότητα και με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλάει με μία φωνή διεθνώς και να προωθεί τα μελήματά της, τα συμφέροντά της με θετικό τρόπο, στραμμένη προς το μέλλον, τη στιγμή που ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ και χάνονται τα σημεία αναφοράς θα πρέπει να είμαστε ε, και πρωταγωνιστής και παράγων ευημερία, σταθερότητας, ασφάλειας για να προωθούμε την πολυμερή συνεργασία. Ε, επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να προετοιμάσουμε στρατηγικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, πολλές διεθνείς συναντήσεις του χρόνου. Έχουμε σημαντικές συνόδους κορυφής με άλλες χώρες ή περιφέρειες του πλανήτη, πρώτα απ' όλα με την Αφρική. Κατά την άποψή μου η Αφρική είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της Ευρώπης και ελπίζω ε, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνουμε μια καλή προετοιμασία για συνεργασία και εταιρική σχέση με την Αφρική και να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Άλλη σημαντική σύνοδος κορυφής του χρόνου, η Κίνα Μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με αυτό το σημαντικό μας εταίρο που είναι η Κίνα και σημαντική χώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ε, συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και καλύτερα για να προωθούμε πάντα και το κοινό μας συμφέρον. Έχουμε στρατηγική σχέση και με τις χώρες αυτές και με άλλες χώρες του κόσμου. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, κλείνω με αυτή τη μικρή εισαγωγή μου λέγοντας το εξή. Τώρα ξεκινάει ένας καινούριο θεσμικός κύκλος. Πιστεύω βαθύτατα ότι ο νέος αυτός θεσμικός κύκλος ε, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Έχουν περάσει λίγο περισσότερο από 60 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης, από τότε που οι πατέρες ίδρυσαν την Ευρώπη, από τότε που κινητοποιήθηκαν οραματιστές, ο Χέλμουτ Κόλ, ο Φρανσουά Μιτερά, που οραματίστηκαν την ελεύθερη κυκλοφορία και το χώρο Σέγγεν, που οραματίστηκαν το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, που αγωνίστηκαν για να προχωρήσει η αλληλοκατανόηση, η ευημερία, η σταθερότητα. Η δική μας πολιτική γενιά, αυτή που και εσείς εκπροσωπείτε στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η δική μας πολιτική γενιά έχει ραντεβού με το μέλλον του ευρωπαϊκού οράματος και εγχειρήματο. Τρεις είναι οι λέξεις που με οθούν. Φιλοδοξία. Φιλοδοξία για τους Ευρωπαίους πολίτες, φιλοδοξία για να μεταφέρουμε αυτό το αισιόδοξο όραμα, εμπιστοσύνη ε, καθημερινή συνεργασία για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων, αλλά κυρίω μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Εμπιστοσύνη στο σχέδιό μα, στις ευρωπαϊκέ αξίε, ε, στο ρεαλισμό, στην κοινή λογική. Ε, να είμαστε προσγειωμένοι και με τα δύο πόδια στην πραγματικότητα, κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη, που έχει και μεγάλες ελπίδες και μεγάλα όνειρα. Το κοινοβούλιο σα είναι καρδιά ίδια της Ευρώπης, μια καρδιά που πάλεται και εκπροσωπείται τα οράματα, τις ελπίδες, τα όνειρα, καμιά φορά και την οργή των ευρωπαϊκών λαών. Τίνω λοιπόν μια χείρα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να συνεργαστούμε για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Μισελ. Πρόεδρε Φοντερ Λάιεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς να συγχαρώ τον πρόεδρο Σαρ Μισελ που προέδρευσε στο πρώτο του Συμβούλιο. Ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή αρχή για την θητεία του. Μια εβδομάδα πριν συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Την επόμενη έφερα την ίδια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο προσυπέγραψε το στόχο να κάνουμε την Ήπειρό μας ουδέτερη κλιματικά μέχρι το 2050. Έχω εξηγήσει στους ηγέτες ε, το, την καρδιά της πρότασής μας, δηλαδή να μεταμορφώσουμε την στρατηγική ανάπτυξη της Υπήρου μας. Διότι για πάρα πολύ καιρό είχαμε αρπακτικές διαθέσεις. Η ανθρωπότητα έπαιρνε πόρους από το περιβάλλον και ως αντάλλαγμα παρήγαγε απόβλητα και ρήπανση. Αυτό πρέπει να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα έχουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα δώσει πίσω στον πλανήτη μας περισσότερα από όσα του έχει πάρει. Μάλιστα, η ηγεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και μία ισχυρή καινοτόμα βιομηχανική βάση πρέπει να θεωρηθούν οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια καθαρή καινοτομία θα χρειαστούμε μακρόπνοες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αλλά αυτή αυτά ήταν πάντα στην καρδιά της ευρωπαϊκής κοινωνικής, ε, ε, ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας της αγοράς, της κοινωνικής οικονομίας. Αυτή λοιπόν η ανταγωνιστική βιωσιμότητα πρέπει να είναι η αρχή μας για το μέλλον στην Ευρώπη. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές αφετηρίες και ειδικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Όπως είπε και ο Σαρλ Μισελ, θα πρέπει να μεταμορφώσουμε σε πολλές περιοχές, περιοχές όπου ε, ως τώρα ζούσαν ανθρακορίχοι, όπως την Ανατολική Γερμανία, ε, σε κάτι διαφορετικό. Ε, κοιτάμε την πρόταση, η Πολωνία ζήτησε περισσότερο χρόνο να δει την πρόταση για τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Ε, έχουμε ήδη αρχίσει να συζητούμε πώς θα υποστηρίξουμε τους ανθρώπους, ε, τις εταιρείες και τις περιφέρειες. Άλλα κράτη-μέλη έχουν άλλα ζητήματα, όπως η Πορτογαλία, που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε δει κυκλώνες, πλημμύρες, ε, τρομακτικές δασικές πυρκαγιές Πέρυσι 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Η Πορτογαλία ξεκίνησε ήδη το 2005 την καθαρή μετάβαση και έχει επενδύσει σημαντικά από τότε. Θα κλείσει το τελευταίο της ανθρακοριχείο το 2023. Ήδη έχει πλεόνασμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μαζί με την κυβέρνηση της Ολλανδίας αυτή τη στιγμή συνεργάζονται για να πετύχουν την πράσινη ενέργεια από το υδρογόνο. Το θέμα είναι πώς ε, η Πορτογαλία θα μεταφέρει τις ανανεώσιμες ενέργειες ε, μέσω της Ισπανίας και της Γαλλίας σε άλλες χώρες που το χρειάζονται. Από την πλευρά των Πορτογάλων η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει να κάνει με τις υποδομές ε, για την ενέργεια, την αλληλοσύνδεση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τρίτο παράδειγμα, η Σουηδία οι εταιρείε ε, χάλιβα αυτή τη στιγμή εργάζονται στο να έχουν παραγωγή χωρίς ε, εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ακούγεται σορεαλιστικό, αλλά είναι χωρί άνθρακα. Είναι επεπισμένοι ότι θα το καταφέρουν σε λίγα χρόνια μάλιστα. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται τη διασφάλιση ότι δεν θα αντιμετωπίσουν το ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Θέλουν η παραγωγή χάλιβα να είναι βιώσιμη για το περιβάλλον και θέλουν να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά χάλιβα. Αυτό και είναι η ουσία της ε, ανταγωνιστικής βιωσιμότητας. Μάλιστα, πολλά από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ζητήσανε για έναν μηχανισμό συνόρων άνθρακα. Το εξετάζουμε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό για να προστατέψουμε τις επιχειρήσεις μας το περιβάλλον και να σεβόμαστε και τους κανόνες του ΠΟΕ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινήσαμε την δουλειά μας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εργασία πριν από πέντε μήνες, εδώ, σε αυτό το ημικύκλιο. Στις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε δώσει σάρκα και οστά στο σχέδιό μας. Το Συμβούλιο έχει προσυπογράψει την συμφωνία. Ε, το δικό σας ψήφισμα μας έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Αυτό που μας περιμένει όμως ως εγχείρισμα είναι τεράστιο. Ε, αν όμως μείνουμε ενωμένοι ως τρία θεσμικά όργανα, ως μία ομάδα, θα κερδίσουμε τη μάχη. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα πόση ισχύ υπάρχει, ε, πόση ισχύς υπάρχει αν είμαστε ενωμένα τα τρία θεσμικά όργανα. Αξιότιμη ευρωβουλευτές, ε, η ευρωπαϊκή φιλοδοξία ε, έχει ανάγκη ε, τις απαραίτητες, τους απαραίτητους πόρους για να πετύχει. Αυτό είναι στην καρδιά της συζήτησης για τον επόμενο προϋπολογισμό. υπάρχουν βέβαια προτάσεις αυτή τη στιγμή που δεν Είναι μακριά από το να πετύχουν αυτό τον στόχο. Ο πρόεδρος Σαρ ε, έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προσπάθειές του να βρει μια ισορροπημένη συνένεση που θα είναι ισότιμη και φιλόδοξη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νταβίτ Σασόλη, που πραγματικά με κάθε δύναμη υπερασπίστηκε ε, τον προϋπολογισμό και με μια ενιαία φωνή. Τον ευχαριστούμε πολύ που το έκανε αυτό στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στις φιλοδοξίες και τις δεσμεύσεις μας. Υπάρχει η στρατηγική ατζέντα του Συμβουλίου, υπάρχουν οι πολιτικές κατευθύνσεις της Κομισιόν και οι δύο προτάσεις ε, είναι συναφείς. Πρέπει όμως για να βρούμε αποτελέσματα, να δούμε αποτελέσματα, να σταθούμε στο ύψος των φιλοδοξιών μας και μας χρειάζονται οι απαραίτητοι πόροι. Αν είναι πολύ μικρός ο προϋπολογισμός δεν υπάρχει παρά μία μόνο λύση. Να συζητήσουμε νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώ που ανέφερες Σαρλ Μισελ το ETS, το Σύστημα Ανταλλαγής Εκπομπών. Είναι και αυτό ε, μία από τις πήγες που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ίδιους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης μιλήσαμε για το διεθνή ρόλο του ευρώ. Το ευρώ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της κυριαρχίας της Ευρώπης στον κόσμο. Όμως ε, ε, είμαστε μία από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, αλλά πρέπει να δούμε ότι πουλάμε το ευρώ μας κάτω από την αξία του. Και εμείς πρέπει να το πετύχουμε, εμείς το έχουμε στο χέρι μας. Θέλουμε ένα κοινό νόμισμα και έχουμε και μια κοινή αγορά από την οποία ε, υποφελούμαστε. Όμως ε, ε, θα πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι να έχουμε και τις διαρθρωτικές προϋποθέσεις για, για ένα κοινό νόμισμα. Αυτό σημαίνει να έρθουμε ένας πιο κοντά στον άλλον. Η Ένωση Κεφαλαίων ε, πρέπει να ολοκληρωθεί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει επιτέλους ε, να επωφεληθούν, να έχουν πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων. Και επίσης η διασυνοριακή δημιουργία, αλυσίδα δημιουργίας αξιών θα υποφεληθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κοινή αγορά και χρειαζόμαστε και την ένωση την τραπεζική. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Ε, δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη κρίση ε, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ε, ανθεκτικότητα του νομίσματός μας. Χαίρομαι λοιπόν που θα έχουμε το λεγόμενο BIC, το ε, δημοσιονομικό εργαλείο για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα, το οποίο έχει κάνει σημαντικές προόδους. Έχουν τεθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του, υπάρχει πολιτική συνένεση για να τεθούν και τα νομοθετικά ε, στοιχεία του και αυτό το μέσο θα οδηγήσει σε μια αλλαγή του τρόπου της εργασίας του Eurogroup θα, βελτιώσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις γιατί ακόμα βέβαια μας λείπει ένα εργαλείο σταθεροποίησης. Υπάρχει λοιπόν το ΣΟΥΡ που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις ασύμετρες ε, εξωτερικές κρούσεις. Μας ε, προστατεύει, προστατεύει την εξειδικευμένη εργασία και αφαιρεί από τις ε, επιχειρήσεις το βάρος. Επίσης δημιουργεί προϋποθέσεις για διαβίου μάθηση και ε, περαιτέρω κατάρτιση. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ξεκάθαρη ε, μια τελευταία λέξη για τον Brexit. Με την ξεκάθαρη νίκη των συντηρητικών και του Μπόρις Τζόνσον, ε, υποθέτω τώρα ότι η συμφωνία αποχώρησης θα κυρωθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Εδώ, σε αυτό το ημικύκλιο, αν κοιτάξω γύρω και κοιτάξω τους ε, βουλευτές, τους γενναίους βουλευτές του Remain. Το μόνο που μπορώ να πω είναι λυπάμαι, θα μας λείψετε. Σας ευχαριστώ για το θάρρος σας. Σας ευχαριστώ που σταθήκατε στο πλευρό μας. We'll Βέβαια αυτούς που φωνάζουν και χτυπιούνται δεν θα, τους, δεν θα μας λείψουν, πραγματικά. και χωρίς εσάς, δόξα το Θεό, θα οικοδομήσουμε τη μελλοντική μας σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σχέση μας πρέπει να είναι όσο πιο στενή γίνεται για το καλό των επιχειρήσεων, των φοιτητών και τόσων Ευρωπαίων που η ζωή τους μοιράζεται στις δύο πλευρές ε, των στενών της μάχης η νέα μας σχέση θα είναι τελείως διαφορετική γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μια τρίτη χώρα. Να ευχαριστήσω τον Μισελ Μπαρνιέ που στο Συμβούλιο και σε όλες τις ε, πλευρές κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων και βοήθησε ε, σε αυτές τις ε, προσπάθειες. Σε ευχαριστούμε. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας είναι γεμάτο προκλήσεις. Πρέπει να έχουμε συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2020 και αν δεν γίνει αυτό θα είμαστε και πάλι στην άκρη του γκρεμού. Αυτό θα βλάψει ξεκάθαρα τα δικά μας συμφέροντα, αλλά περισσότερο θα έχει αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να επωφελείται από την ενιαία αγορά, από την Τελωνιακή Ένωση και από τις 750 διεθνείς συμφωνίες που έχει συνήψει με τους εταίρους της. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν είναι προς συμφέρον μας να μην υπάρχει τέτοια συμφωνία. Θέλουμε λοιπόν να οργανώσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, για να, να έχουμε αποτελέσματα όσο πιο σύντομα γίνεται και να έχουμε και ένα, μια θητεία στην 1η Φεβρουαρίου. Θέλουμε ε, να ξέρουμε πια ότι ε, με την Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα η εταιρική μας σχέση θα είναι καλή. Δεν θα είναι το τέλος. Θα είναι η αρχή νέων σχέσεων μεταξύ γειτόνων. Και θέλω πραγματικά να γίνουμε καλοί γείτονες με τους φίλους μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζήτω η Ευρώπη. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Φόντε Και τώρα λόγο στον Πρόεδρο Βέμπερ. Παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έρχεστε πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβετε καθήκοντα και να μιλήσετε στο σώμα μας. Βεβαίω ε, και με τα προηγούμενα καθήκοντά σα και επειδή είστε από το Βέλγιο, είστε γνώστη ε, τη πολιτική. Ε, θα χρειαστείτε πολύ τύχη βέβαια και για τα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, είναι ένα θεσμικό όργανο που μπλοκάρει τι αποφάσει. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και τι επόμενε εβδομάδε, διότι θα πρέπει να δούμε και τις επιτυχίες που θέλουμε να πετύχουμε για το κλίμα ως 27 και πώς μπορούμε να καλύψουμε το κόστος για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Ε, θα πρέπει να γίνει εδώ μια σημαντική συζήτηση. Η Φινλανδική Προεδρία ε, θα πρέπει να οργανώσει συζητήσει, ε, οργάνωσε συζητήσει με επιχειρηματίε ε, και θα πρέπει να συμμετέχουν πλέον όλοι επιχειρηματίε, φοιτητέ, ε, πολίτε. Αυτό το ζήτημα δεν μπορούμε πλέον να το αποφεύγουμε. Έχουμε λοιπόν μεγάλες ευθύνες να λάβουμε και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι σχετικές συζητήσεις αμέσως. Επίση, μεταξύ των επιτυχιών τη Φιλανδικής Προεδρίας, για μας, με τις προτάσεις που είδαμε από τη Φιλανδική Προεδρία, είχαμε μια απλή πρόκληση. Διότι δεν είναι ο προπολογισμό που προτάθηκε αρκετό για τι επενδύσει που χρειάζεται στο μέλλον η Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρξει μελλοντικά μια συζήτηση για το ποιε θα είναι οι αρμοδιότητε που θέλουμε να φέρουμε πέρα. Ποιο θα πληρώνει και Όταν ε, η χώρα μου, η Γερμανία, προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα χωρών η Ιταλία και η Ελλάδα, αυτό είναι ένα όφελος κοινό και για, την, ε, για τους Γερμανούς Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ε, στο δεύτερο, θα πρέπει να, το δεύτερο θέμα στο οποίο να δώσουμε προσοχή είναι ότι θα χρειαστούν συζητήσεις με τόλμη το επόμενο, τα επόμενα χρόνια. Το κράτος δικαίου, κάτι που έχει απασχολήσει ήδη το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Ρουμανία. Ε, υπάρχουν ε, θέματα για το μέλλον, διότι υπάρχει καταστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εβδομάδα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο θα συζητήσουμε για τη Μάλτα. Νέα δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε γιατί απλώς έκανα τη δουλειά της και αυτό επειδή η ελίτ ε, του κράτους ήταν διεφθαρμένη. Ε, ο Πρωθυπουργό μπορεί να έχει ευθύνε. Υπήρχαν ε, επαφές μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και πολιτικών. Αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο Συμβούλιο. Δεν μπορεί να αποσιωπάται. Δεν μπορεί να είναι αυτό κάτι που να επιτρέπεται σε Ευρωπαίους ηγέτες. Θα πρέπει θέματα όπω η Ουγγαρία, η Δημοκρατία τη Τσεχία, η Πολωνία, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει να έχουν το θάρρο να μιλήσουν με αυτού του συναδέλφου του, του ομολόγου του. Ε, συνάδελφοι, ω ΕΛΚ θα πρέπει επίση να δούμε και την πραγματικότητα του Brexit. Ε, ξέρουμε τι εντολή έχει αναλάβει ο Μπόρι Τζόνσον και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Κίφερ Χόφστατ για τη δουλειά που έκανε εκ μέρου του Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει από την πλευρά μα ό,τι μπορούσαμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με την μελλοντική συμφωνία και θα πρέπει να βασιστούμε σε μια φιλική σχέση για τη μελλοντική μας ακριβώς ε, ε, σχέση. οι περισσότεροι Βρετανοί θέλουν μια ισχυρή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να φροντίσουμε για τα συμφέροντα όλων μας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να γίνονται ε, δεκτοί και οι κανόνες για την αγορά μας, όπως, θα πρέπει να, όπως πρέπει να ισχύουν και για το σύντη του Λονδίνου και για τα προϊόντα. Και εκεί θα πρέπει να βασιστούμε για τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει όπου θα παίξει ένα ρόλο και το Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εταιρική σχέση που θα πρέπει να δούμε πώς θα καθορίσει την μελλοντική σχέση γειτονίας που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Και επίσης για το τελευταίο, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και το πόσο μπορούν να ανοίξουν οι διαπραγματεύσει με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Περιοχές που έχουν γνωρίσει μεγάλη απογοήτευση με την πρόσφατότερη απόφαση. Εδώ μετά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σας ζητούμε ως ΕΛΚ να σκεφτείτε το θέμα των διαπραγματεύσεων ε, με αυτέ τι δύο χώρε. Θα πρέπει να το δούμε και μελλοντικά και να ξεκινήσει η διαδικασία προσχώρησής του. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Γκαρσία Πέρε. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Γκαρσία Πέρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Αγαπητέ κύριε Μισελ, εξ ονόματο της ομάδας μου σας καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε η Προεδρία σας να αποδειχθεί ισχυρή και ηγετική για να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα και τις προκλήσει στην Ευρώπη. Θάρρο χρειάζεται στη λήψη των αποφάσεων και ηγετική στάση. Είμαστε υπεύθυνοι για τι δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε σε όλε τι συζητήσει που γίνονται στο Συμβούλιο. Αν φιλοδοξούμε να έχουμε μια Ευρώπη πιο οικολογική και χωρί αποκλεισμού και πιο κοινωνική, χρειαζόμαστε χρήματα που να είναι στο ύψο των φιλοδοξιών μα Και επίση χρειαζόμαστε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο στιβαρό και γερό για να αντιμετωπίσει η μελλοντική οικονομική κρίση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών μα, ανδρών και γυναικών, στα πλαίσια μια πολιτική κοινή, εξωτερική και πολιτική ασφάλεια. Αξιολογούμε θετικά το γεγονό ότι το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, παρά την αντίσταση κάποιου κράτους μέλους. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε όταν συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης. Ότι χρειάζεται να αλλάξει ο κανόνας της ομοφωνίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρούμε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε. Παρόλο που τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ήταν ένα ταμπού που δεν συζήτησε κανείς. Οι περικοπές αυτές είναι τελείως απαράδεκτες. Η ομάδα μας περιμένει να αλλάξει αυτό ε, το πλαίσιο. Η τωρινή πρόταση του Συμβουλίου είναι τελείως ανεδαφική. Λιγότερα χρήματα για τη συνοχή, λιγότερα χρήματα για τη γεωργία, λιγότερα χρήματα για τη διασύνδεση της Ευρώπης και τη διαχείριση των συνόρων. Και αναφέρω επιγραμματικά μόνο μερικά θέματα. Επίσης, ε, είναι ανεπαρκής η χρηματοδότηση της πρότασης για την πολιτική της έρευνας και για τους κλιματικούς στόχους. Και κάτι που είναι ακόμα χειρότερο, δεν γίνεται πουθενά αναφορά στο Ταμείο Δίκαιης μετάβασης και ε, στην εγγύηση για τα παιδιά ε, και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες με λιγότερη χρηματοδότηση. Αν δεν θέλουμε να μείνει κανείς πίσω, θα πρέπει το Συμβούλιο να ποντάρει σε ένα ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό από επιπλέον ιδίου πόρου και εθνική ε, επένδυση. Γι' αυτό θέλουμε να μπει ο Χρυσό κανόνας ε, στο Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, έτσι ώστε να μην υπολογίζονται οι επενδύσεις για την πράσινη οικονομία ε, ως επενδύσεις που επιβαρύνουν τους προπολογισμού. Θα πρέπει επίσης ο κοινωνικός πυλώνας να μπει στο εξάμεινο το ευρωπαϊκό και να μην είναι απλώς συμβολικό αυτό. Ε, ε, θα πρέπει να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια και να συνδέονται ε, με τον κοινωνικό πυλώντα τα διαρθρωτικά ταμεία. Κύριε Μισελ, αν θέλουμε να επιτύχουμε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι και παιδαγωγία και ενσυναίσθηση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κατανοούν το ένα το άλλο και να διαπαιδαγωγούν τους πολίτες. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο ευεργετικό να είναι πιο ισχυρή Ένωση. Και για το Brexit, τελειώνω. Σήμερα θα μου επιτρέψετε επευκαιρία να στείλω ένα σαφές μήνυμα αναγνώρισης και ευχαριστειών προς τους ευρωβουλευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο που επί 46 έτη έγραψαν ιστορία εδώ στη δημοκρατία μας, στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Προηγουμένως συζητούσαμε τη δέκατη επέτειο της Λισαβόνας. Ο συνάδελφός μας Ρίτσαρτ Κόρμπετ ήταν εισηγητής για τη συνθήκη αυτή. Αξίζεται το σεβασμό μας, αξίζεται την αναγνώρισή μας, αξίζεται επίσης την αγάπη μας και την προσωπική. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Κανείς δεν πρόκειται να σας αφαιρέσει την υπερηφάνεια αυτή ε, που είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε στην ιστορία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Σας ευχαριστώ όλους και όλους σας. Ευχαριστούμε πρόεδρε Τσόλος. Euh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Σαλ, καταρχά, ε, να σα συγχαρώ για την ανάληψη των ε, αυτής ε, της θέσης ε, έχουμε να αποθέσει πολλές ελπίδες ε, στην έναρξη αυτής της θητείας γιατί έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα πραγματικό εταίρο ο οποίος θα μπορέσει να προωθήσει τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Στις τελευταίες ευρωεκλογέ το μήνυμα των πολιτών ήταν ξεκάθαρο. Τώρα σε εμά αναπόκειται να εφαρμόσουμε όλα αυτά. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι εσύ έχεις το όραμα, έχεις τη δυνατότητα να φέρεις εις πέρας τις διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε όσα χρειάζονται για να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αυτό το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο προείδρευσες μας έφερε καλά νέα με τις δεσμεύσεις ε, για το κλίμα μέχρι, μέσα στον ορίζοντα που έχουμε μέχρι το 2050. Υπάρχουν στο Συμβούλιο βέβαια πολλά κράτη-μέλη που ακόμα μπλοκάρουν και ακόμα δεν υπάρχει κατάλληλη αποφασιστικότητα για να εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι. Γιατί εντάξει, καλό να υπάρχουν στόχοι και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά ήδη, όμως τώρα πρέπει να μπορούμε και να τους εφαρμόσουμε. Και γι' αυτό ε, πρέπει η Κομισιόν να έρθει με προτάσεις. Χρειαζόμαστε να δώσουμε το θάρρος στα κράτη-μέλη να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και να κάνουν αυτό το βήμα μπρος. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρέπει να μεταμορφώσουμε αυτό αυτό το εγχείρημα για το κλίμα σε μια ευκαιρία. Υπάρχουν βέβαια κάποια κράτη-μέλη που ξεκινούν από διαφορετικά σημεία, είναι άλλη αφετηρία τους, όμως ε, είναι πραγματική ευκαιρία η προσπάθεια αυτή κατά της κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά πρέπει να τα μεταφράσουμε και στις δημοσιονομικές προοπτικές για να μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα όχι μόνο σε επίπεδο περιβάλλοντος αλλά και στην ψηφια... στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε όλους τους στόχους. Το πολιτές μου δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να είναι ένα πραγματικό εργαλείο για την Ευρώπη. Όχι μόνο μια διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών ε, μελών που δίνει ε, κέρδη στους μεν ε, και χασούρα στους δε. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, αν το δούμε έτσι, θα είναι και ο μόνος τρόπος να έχουμε μια σωστή απόφαση για τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Να κατανοήσουμε δηλαδή ότι το ΠΔΔ είναι ε, ένα εργαλείο για τις φιλοδοξίες μας, όχι για παζάρια στα οποία κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν για τις δημοσιονομικές προοπτικές κατά τη γνώμη μου θα ήταν λάθος να μετράμε πόσα δίνουμε στις κλασικές πολιτικές, τις παλιές και πόσα βάζουμε στις νέες προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε έναν εξυγχρονισμό. Οι κλασικές πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική συνοχής χρειάζονται μεταρρύθμιση για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στις τρέχουσες ανάγκες και να μην εξασθενούν τις δυνάμεις της Ένωσης. Ε, ε, επίσης, ε, υποστηρίζουμε έναν ισχυρό προϋπολογισμό γιατί ε, πραγματικά πρέπει να γίνουν ε, σημαντικά βήματα μπρος. Ε, χρειαζόμαστε να αλλάξουμε τη στάση μας ως προς τους ίδιους πόρους. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία όλη την ώρα μιλάνε για το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Οι ίδιοι πόροι είναι ένα πρώτο βήμα για να έχουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο θα είναι δομημένος με βάση ευρωπαϊκούς στόχους και προθέσεις. Τέλος, ε, μια λέξη για το Brexit. Λυπόμαστε για τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τουλάχιστον όμως τώρα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι θα συμβεί. Το Κοινοβούλιο θα αναλάβει την ευθύνη του. Θα ήθελα όμως επίσης να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πίστεψαν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, που μετέδωσαν ξεκάθαρο μήνυμα στους Βρετανούς ότι το Brexit δεν είναι το τέλος της κοινή μα ιστορίας και ότι θα παραμείνουμε εταίροι. Ε, θα είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι όλοι οι Βρετανοί που πραγματικά πιστεύουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα θα μείνουν ενωμένοι μαζί μας και θα βρούμε το σωστό τρόπο να συνεργαστούμε και να εργαστούμε από κοινού. Ευχαριστούμε τον Μισελ Μπαρνιέ και τον Γκίφερ Φερχοφστατ για τα όσα έκαναν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να έχουμε μια καλή και ισχυρή συμφωνία με τους γειτόνους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Κέλλερ. Παρακαλώ Σκα. Συνάδελφοι, ενώ η Αρχηγή Κρατών και Κυβερνήσεων συναντιόταν στη Βρυξέλλε την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε η COP25 στη Μαδρίτη που καθυστερούσε ε, και τελμάτωνε. Θα ήταν ε, πολύ καλή ιδέα του χρόνου στην Γλασκόβη, στην COP26, ε, όχι όπως στη Μαδρίτη, επιτέλους να δείξουμε τη σημασία που θέλουμε να αποδώσουμε στη συναντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, ιδίως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνεδρίαζαν ταυτόχρονα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τους στόχους μας μέχρι το 2050, όπως συζητήθηκαν στη διάσκεψη και τη μείωση μέχρι 30%. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στόχο, αλλά το 2050 είναι πάρα πολύ αργά ούτω ή άλλω. Και η θέση στόχων είναι μόνο το μισό από αυτό που έχουμε να κάνουμε. Η πραγματική μα μάχη δεν είναι απλώ η μελλοντική στόχη. Αυτό που μετράει είναι τι δράσει θα αναλάβουμε σήμερα, προκειμένου να πετύχουμε του στόχου αυτού. Για τι συγκεκριμένε λοιπόν ενέργειε που χρειάζονται, πρέπει να δούμε το ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, το μακροχρόνιο προπολογισμό μα, δηλαδή το ευρωπαϊκό προπολογισμό Πρέπει να υποστηρίζει την επίτευξη των κλιματικών μα στόχων, όχι να του υπονομεύει. Και αυτή τη στιγμή οι προτάσει που έχουμε επιτάπητο δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων. Δεν καταφέρνουν να φτάσουν εκεί που πρέπει για το κλίμα. Και πολλέ επιδοτήσει δεν έχουν καλυφθεί, πολλέ δεν έχουν καθόλου στόχο την προστασία από το, κλιματικέ κλιματικές αλλαγές και την προστασία τη βιοποικιλότητα. Ελπίζω λοιπόν τα κρατημέλη να αρχίσουν να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά για το κλίμα και τον προπολογισμό. Και ε, είδαμε ότι η πολωνική κυβέρνηση απομονώθηκε δεν συμφώνησε με το στόχο. Ε, να μην ξεχνάμε ότι 70% των Πολωνών των ίδιων είναι υπέρ των στόχων αυτών. Οπότε η πολιτική κυβέρνηση καλό θα ήταν να αλλάξει γνώμη. Διότι όσο πιο αργά ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση, τόσο πιο δύσκολη θα είναι. Γιατί οι κλιματικέ αλλαγέ δεν σταματάνε στα σύνορα καμιά χώρα. Brexit. Το Brexit είναι και παραμένει μια τραγική υπόθεση. Βεβαίως, δεν είναι το τέλος. Δεν θα τα παρατήσουμε. Ποτέ δεν θα παρατήσουμε τους Βρετανούς φίλους μας. Δεν θα τους ξεχάσουμε. Και ποιο ξέρει, ίσως μια μέρα να μπορούμε να πούμε «Καλώς ήρθατε και πάλι, Ηνωμένο Βασίλειο. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σα. Ευχαριστώ κύριο Άνεμαντς. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πολλοί στο Βέλγιο και πολλοί στη Βλάνδρα θυμούνται τον Νάιτζελ Φαράντς πώς είχε καλωσορίσει τον προηγούμενο ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, θα σας χαλάσω λίγο το πάρτι εδώ πέρα που χαίρεστε και καλωσορίζετε. Ακούσαμε τον κύριο Μακρόν για το Σπίτσεν Καντιντά, το κορυφαίο υποψήφιο που σας τα χάλασε ε, και ε, ε, βασικά για να επιλέξουν κάποιο υποψήφιο έπρεπε να είναι γαλλόφωνος και πήραν κάποιον από το Renew Europe γαλλόφωνο και τον βάλανε πρόεδρο του Συμβουλίου. Το Βέλγιο είναι μια ε, περίπλοκη χώρα και είπανε ας πάρουν ένα Βέλγο πρωθυπουργό θα είναι καλός μάνατζερ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και πάλι λάθος κάνατε. Είναι από τα χειρότερα κράτη-μέλη το Βέλγιο ο προπολογισμό μας. Χάρη στον κύριο Μισελ. Έχουμε 11 δισεκατομμύρια ε, Είμαστε κοντά στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μην νομίζετε, είναι ψευδέστηση ότι το Βέλγιο ε, είναι μια χώρα με καλή διαχείριση. Ούτε οι πολίτες του Βελγίου δεν το πιστεύουν αυτό. Ε, Χτες κλείσαμε 365 ε, μέρες κυβερνητικής κρίσης στο Βέλγιο και κανένας από την πολιτική ελίτ του Βελγίου δεν ξέρει τι κυβέρνηση θα έχουμε. Κάναμε και εκλογές και τώρα κάνουμε ανάλυση ε, ε, ότι χρειάζονται και νέες εκλογές. Δεν μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση αυτή η χώρα. Ε, στο μεταξύ, κυβερνάνε τα, τα απομεινάρια της κυβέρνησης ε, Μισελ. Έχει 38 βουλευτές από τους 150. Είναι μια χώρα που κυβερνάει η μειοψηφία με τρόπο δικτατορικό. Και μιλάτε και για πολυμερή συνεργασία. Εδώ δεν μπορείτε να έχετε κυβέρνηση στη χώρα. και με μαζική μετανάστευση. Και ε, έριξε την κυβέρνησή του ε, γιατί ήθελε να πάει στο Μαρακές να υπογράψει το σύμφωνο ε, για τη μετανάστευση. Λοιπόν, αγαπητοί πολίτες, μιλώ στα αγγλικά τώρα και ως πολίτης που ζω στο Βέλγιο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο λεγόμενος πρόεδρος σας του Συμβουλίου δεν είναι νοτικός, αλλά είναι μάλλον πηγή πολιτικού χάου και θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Εμεί τη ομάδα ID είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής συνεργασίας αλλά στεναρά κατά του όλο και πιο στενού ευρωπαϊκού κράτου. Ελπίζουμε ο Σαρ Μισελ να αποδειχθεί τόσο καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αποδείχθηκε για το Βέλγιο. Ο κύριος παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, το Συμβούλιο συζήτησε πολλά σημαντικά θέματα την τελευταία εβδομάδα, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ στο Brexit. Οι συντηρητικοί όντως ε, ε, είχαν μια ιστορική νίκη την περασμένη Πέμπτη. 365 είναι τα μέλη του συντηρητικά του Κοινοβουλίου, είναι 80 πάνω από τα υπόλοιπα ε, κόμματα. Ήταν πάνω από όλα όμως μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνη στον Μπόρις Τζόνσον ως Πρωθυπουργό. Ε, για να πήρε και την εντολή να ολοκληρώσει το Brexit. Επίσης ήταν πλήρης απόρριψη ε, του σοσιαλισμού με τον τρόπο που τον πρόσφερε το εργατικό, το εργατικό κόμμα. Δεν ε, θα επιτρέπεται πλέον στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπαίνουν στα εδάφη μας και να ε, περνά, ε, να κραδένουν τις σημαίες, τις μπλε σημαίες ή να έρχονται σε μας ε, και να στέλνουν λάθος μηνύματα που οδηγούν σε παρεστήσεις. Το, Ευρωπαϊκό, η Ευρω... το Βασίλειο θα προχωρήσει σε μια ευέλικτη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και άλλους τομείς συνεργασίας για να μπορέσουμε εκ να φτιάξουμε μια νέα σχέση φίλων κυρίαρχων ισότιμων κρατών. Αυτή είναι μια πρόκληση, είναι το μεγάλο εγχείρημα του 2020 που τροφοδοτήθηκε με τις πιο θερμές ευχές ε, του, Προέδρου μας για, ε, του Πρωθυπουργού μας για τα άλλα ε, κράτη. Ευχαριστώ την Πρόεδρο Φοντερ Λάιεν για τις θετικές παρατηρήσεις της και όλα τα υπόλοιπα μέλη γιατί πραγματικά θα πρέπει τώρα να βιαστούμε για την συμφωνία. Θα ψηφιστούν όλα αυτά στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας και ε, θα φύγουμε την 31η Ιανουαρίου. Έτσι, με καλή πίστη θα έχουμε ταχεία πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική μας σχέση για να έχουμε μια καλή ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ε, που θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη του 2020. Αυτό πρέπει να είναι και ο κοινό μας στόχος. Ξέρω το Μισελ Μπαρνιέ προσεγγίζει όλα αυτά τα θέματα με θετικό πνεύμα και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχουμε τις προθεσμίες. Ευχαριστώ λοιπόν το Σώμα και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μισελ, σας καλωσορίζω στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η πρώτη σας παρουσία εδώ. Η πολιτική μου ομάδα έχει μεγάλες διαφορές με την πολιτική σας, αλλά ομολογώ ότι η σκληρή επίθεση που δέχεστε από την ακροδεξιά εδώ μέσα στο ευρωκοινοβούλιο ε, ανεβάζει και τον πύχη των προσδοκιών που έχουμε από εσά. Και θέλω να πω ότι το πρώτο πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι να πάψει το Συμβούλιο να μπλοκάρει πράγματα που ζητά το Ευρωκοινοβούλιο, απαιτούν οι καιροί και ορισμένα από αυτά τα στηρίζει και η Κομισιόν. Και σταματούν στο Συμβούλιο. Ξεκινώ από ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ την ομάδα μας αλλά με αφορά πολύ και ως Έλληνα. Δεν αρκεί κύριε Μισελ η φραστική καταδίκη της επιθετικότητας του καθεστώτος Ερντογάν που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, που απειλεί την Κύπρο και την Ελλάδα και που απειλεί να βάλει φωτιά σε μια ευαίσθητη περιοχή. Δεν αρκεί η φραστική καταδίκη απαιτούνται κυρώσεις και το συμβούλιο έχει αποφασίσει κυρώσεις τον ιούνιο και τον οκτώβριο αλλά πρέπει να τις ενεργοποιήσει. θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε γιατί δεν ενεργοποιείτε αυτές τις κυρώσεις. και το δεύτερο για να υλοποιηθούν οι στόχοι που και εσείς παρουσιάσατε και η κυρία φόντερ λάιεν παρουσίασε για την κλιματική αλλαγή για την κοινωνική συνοχή για την αγροτική πολιτική για την τεχνολογική ανανέωση απαιτούνται χρήματα και το ευρωκοινοβούλιο με μια μεγάλη πλειοψηφία έχει καταλήξει σε μια πρόταση που λέει για να υπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι χρειαζόμαστε τουλάχιστον το 1,3% του ευρωπαϊκού αεπ. η δική μου πολιτική ομάδα θα ήθελε και πιο φιλόδοξου στόχου για την κοινωνική ατζέντα για το κλίμα αλλά έστω αυτό που προτείνει το ευρωκοινοβούλιο με μια μεγάλη πλειοψηφία και έρχεται το συμβούλιο δια της φιλανδικής προεδρίας και προτείνει περικοπέ. 13% στην περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, 27% στις επενδύσεις για τον άνθρωπο και την κοινωνική συνοχή, 25% περικοπές για το LIFE, για το κλίμα, 30% στο πρόγραμμα Horizon, 48% στο πρόγραμμα Erasmus σε σχέση με τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, 35% στο πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη. Και την ίδια ώρα, αν συγκρίνουμε τις προτάσεις σας για το νέο πολιετή προϋπολογισμό σε σύγκριση με τον προηγούμενο προτείνετε 132% αύξηση για την μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων και 650% για την στρατιωτικοποίηση, την άμυνα και την ασφάλεια. Ποιον πολίτη μπορείτε να πείστε με αυτή την πολιτική. Και ως πότε θα καθυστερείτε και θα αναβάλλετε αυτό που χρειάζεται. Γιατί αλλιώς όλα τα ωραία πράγματα που ακούστηκαν και από την κυρία Φόντερ Λάιεν και από εσά για την κλιματικά ουδέτερη πολιτική για την κοινωνική ατζέντα για τους αγρότες για την κοινωνική συνοχή θα μείνουν λόγια. σε αυτά θα ήθελα απαντήσει στη δευτερολογία σας. σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ο Ευχαριστώ. Είμαι ένας υπερήφανος Βρετανός σήμερα, γιατί έχουμε κερδίσει τη μάχη για το Brexit. Είμαι περήφανος για τους φίλους μου του κόμματος του Brexit και πραγματικά ε, θα προσπιστούμε τη Βρετανική Δημοκρατία και είμαι υπερήφανος για τον Βρετανικό λαό που πήγε και ψήφισε στις γενικές εκλογές σωστά. Ε, ε, επιστηρίξανε το Leave, την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ότι προσπαθείτε να καλλιεργήσετε ένα μύθο για τους Βρετανούς. Αλλά εμείς δεν σας πιστέψαμε. Και τώρα, επιτέλους, θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία μας, του ε, μεγάλου μας έθνους ε, θα πάρουμε πίσω τους ε, πόρους μας, τα χρήματα, τα, ε, τις, τα προϊόντα μας, τις εταιρείες μας και θα μπορέσουμε να καθορίσουμε εμείς το μέλλον μας. Το μέλλον της Βρετανίας είναι λαμπρό με τον Brexit. Και ε, ε, ελπίζουμε ο Μπόρις Τζόνσον, αυτή είναι η έκκλησή μας προς αυτόν, να μην παραδώσει τα όπλα. Επιτέλους ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω την κατάσταση στα χέρια μας. Ευχαριστούμε κυρία Χίμπνερ για 1,5 λεπτό. Um, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν καλό κάποια μέρα να ακούσουμε που είναι ο πολιτικός σας χώρος. Ε, πού θα πάτε όταν φύγετε από το Κοινοβούλιο. Πρόεδροι, αξιότιμε Μισελ Μπαρνιέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την ε, σαφήνεια που θέλουμε για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και ζητά λοιπόν, βλέπουμε ότι οι φίλοι μας ε, θα γίνουν μια τρίτη χώρα στα τέλη του Ιανουαρίου. Λυπάμαστε γι' αυτό, αλλά το σεβόμαστε. Υπάρχουν φιλίες που θα παραμείνουν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το δικό μας μερίδιο για να οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγκαίρως. Ε, λυπόμαστε που φεύγουν οι φίλοι μας, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Σημειώνουμε τη στρατηγική πρόθεση του ε, Πρωθυπουργού της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Ε, όμως λυπόμαστε που θα έχουμε ε, μπλοκάρει με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν με καλή πίστη. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το μέλλον και αδειμονούμε για επικοδομητικές συζητήσεις, γιατί θέλουμε μια φιλόδοξη συμφωνία. Η εντολή μας θα βασιστεί στις πολιτικές δηλώσεις που το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού συμφώνησαν. Ελπίζουμε ότι η πολιτική δήλωση αυτή ε, θα πάει ε, σε μεγαλύτερο βάθος ε, και θα είναι η πιο βαθιά και πολυπίκυλη συμφωνία που έχουμε με τρίτη χώρα. πρέπει μαζί να ανταμώσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις εδώ σε αυτό το σώμα δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τη σωστή εφαρμογή και, τη σωστή παρακο... και την ε, στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκραπίνη ζητάει μπλε κάρτα. Όμως δυστυχώς ε, ε, πιέζομαι να τελειώσουμε και δεν μπορούμε να πάρουμε μπλε κάρτες. Δεν έχουμε χρόνο, κυρία Γκραπίνη. Έχουμε πρόβλημα και με το Catch the Eye. Δίνω τώρα ε, στην κυρία Μποναφέ το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε εδώ λόγια πολύ σημαντικά από την πλευρά του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίω ε, για την Πράσινη Συμφωνία. Χαιρόμαστε που το Συμβούλιο δεσμεύεται με τα συμπεράσματά του, εκτό τη Πολωνία βεβαίω δυστυχώ, να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έω το 2050 βάσει τη Συμφωνία των Παρισίων. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι καμπή ιστορική σημασία η Πράσινη Συμφωνία. Ε, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα διαβίωση και τι κοινωνικέ συνθήκε στην Ευρώπη. Η Πράσινη Συμφωνία πέτυχε ένα πρώτο αποτέλεσμα, δηλαδή να θυμίσει τι ανάγκε των πολιτών και πραγματική οικονομία πρέπει να έρθουν στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών μετά από χρόνια συζητήσεων που έχουν απασχοληθεί με τι παράμε, παραμέτρου του, δημόσιου, του κρατικού χρέου και των προπολογισμών των δημοσιονομικών στα κράτη-μέλη. Όμω αυτό που σκιάζει την όλη αυτή επιτυχία είναι οι επενδύσει. Δεν είπα τότε μια κουβέντα για αυτό, κύριε Μισελ, και χρειάζονται κινήσει, συγκεκριμένε ενέργειε. Πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση τη Πράσινη Συμφωνία χωρί να στρεφόμαστε γύρω από την ουρά μα. Χρειάζεται ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο στο ύψο των περιστάσεων και των προκλήσεων του μέλλοντο και θα πρέπει να ε, ξαναδούμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, δίνοντα τη δυνατότητα στα κάτι μελη να μετρήσουν στο έπτου του επενδύσει εφόσον αυτέ επιτρέπουν την επιτέξη των στόχων τη Πράσινη Συμφωνία. Η πρόεδρο Φοντερ Λάιν έδειξε τόλμη και αποφασιστικότητα, όμω εάν δεν την στηρίξουν οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων, ε, ο δρόμο τη ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα είναι ανηφορικό και δύσκολο. Ευχαριστούμε κύριε Φερχόφστατ για 2,5 λεπτά. Το πρώτο που θα ήθελα να πω στον κύριο Άνεμαν είναι ότι αυτά που είπαν είναι σκανδαλώδη. Εγώ είμαι περήφανο που ένα Βέλγο είναι πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντί όλε αυτέ τι ανοησίε που είπατε. Και αν δεν γνωρίζετε, συνάδελφοι, για ποιο λόγο υπάρχει μειοψηφία στο Βέλγιο, λόγω των αποσχιστών ε, του κυρίου Άνεμανς. Αυτή είναι η μειονότητα στο Βέλγιο. Και στον κύριο Φαράνς και, και ε, τους δικούς του, θέλω να πω ότι κάνουν πολλή φασαρία εδώ ε, για ε, τις εκλογές. Και όλοι είπαν εδώ ότι θα μας λείψουν οι Βρετανοί συνάδελφοι, ε, οι εργατικοί, οι φιλελεύθεροι. Οι ε, του Brexit δεν θα μου λείψουν καθόλου και σας το λέω. Καθόλου δεν θα μου λείψουν. Εν πάση περιπτώσει αγαπητοί συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει σύμφωνη γνώμη, ξέρετε. Ξέρω όλοι θεωρούν ότι εντάξει αυτά είναι αυτόματα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή η διαδικασία έγκρισης θα έρθει στις 29 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια. Στο μεταξύ πρέπει να λυθεί ένα πρόβλημα όμως. Έχω λάβει από τις εκλογές στη Βρετανία εκατοντάδες εκατοντάδων επιστολών και mail Βρετανών πολιτών που ζουν στην Ευρώπη και είναι πανικόβλητοι για το μέλλον τους και το καθεστώς που θα έχουν. Έχω λάβει εκατοντάδες mail πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στη Βρετανία, οι οποίοι είναι επίσης πανικόβλητοι για το τι θα τους ξημερώσει και νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να λύσουμε αυτά τα προβλήματα πριν δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για τη συνθήκη του Brexit. Για ποιο λόγο αγαπητοί συνάδελφοι, ποτέ οι πολίτες, οι Βρετανοί ή Ευρωπαίοι να είναι θύματα αυτή τη επιλογή που κατά τη γνώμη δεν ήταν και η ευφιέστερη για τον Brexit. Και θέλω να απευθύνω μια έκκληση στον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπόρι Τζόνσον. Να είναι γενναιόδωρος στη νίκη του και να δώσει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο όλα τα δικαιώματά τους, τα πλήρη, τα οποία απολαμβάνουν σήμερα, αυτόματα σε όλους, χωρίς αστερίσκους και χωρίς αλλά, όπως ε, συνηθίζει να λέει και αρέσκεται. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όλο και περισσότεροι επιστρέφουν, και τελειώνω με αυτό, σε ένα άλλο θέμα οι ε, Βρετανοί που θέλουν να εξακολουθούν να είναι Ευρωπαίοι να έχουν κάποιο είδο ευρωπαϊκή ηθαγένεια, συνδεδεμένη ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Ο κύριο Άικχαουτ, 1,5 λεπτό. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, Πρόεδρε Σαρ Μισελ, καλώ ήρθατε και συγχαρητήρια για το πρώτο σα συμβούλιο. Τα συμπεράσματά του ε, σχεδόν ομόφωνα για την κλιματική ουδετερότητα ε, τα λέμε με νομόφωνα, αλλά τέλος πάντων είναι σημαντικά. Και επίσης σημαντική είναι και η συζήτηση που σας αναμένει για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πουδουπού. Ε, εδώ πολλές χώρες συζητούν για τις κλιματικές δράσεις, τις κλιματικές φιλοδοξίες και μεταξύ αυτών και η δική μου ίδια ε, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κλιματικές δράσεις χρειάζονται βεβαίω και κάποια χρηματοδότηση. Πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε σε σχέση με τα κονδύλια και οι κατοχώρες και η Δανία και η Σουηδία και η Αυστρία και η Φινλανδία όταν δεν θα είναι πια προεδρία θα πρέπει να μεταφράσουν αυτές τις φιλοδοξίες τους και σας σε ε, υψηλότερα κονδύλια, μεγαλύτερο προπολογισμό για να μπορέσει να γίνει η μετάβαση για το κλίμα. Δεύτερο σημείο, και αυτή είναι ερώτηση προς εσάς, σας ε, πήρε, τουλάχιστον όχι σε εσάς ειδικά, στο Συμβούλιο, δυόμιση χρόνια για να φτάσετε σε μια συμφωνία για το στόχο στο 2050. Έχουμε μόνο ένα χρόνο μέχρι να πάμε στη Γλασκόβη για να συμφωνήσουμε για το στόχο στο 2030. Ε, στο ενδιάμεσο, το Σεπτέμβριο έχουμε και μια σημαντικότατη σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Πώ να είμαι βέβαιο ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι ε, έτοιμο για καλύτερου, βελτιωμένου στόχου για το 2030 πριν ε, το Σεπτέμβριο στη Λιψία και στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση και ελπίζω να μπορώ να σα συγχαρώ για τα ε, αποτελέσματά σα ω τον Ιούνιο. Ευχαριστούμε κύριε Μπάι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σήμερα ε, παρακολουθούμε το χορό όσων δεν ξέρουν να χάνουν. Σοσιαλιστές, Γκίφερ Χόφστατ λυπούνται για τη δημοκρατική επιλογή του Βρετανικού λαού. Η ετοιμιγορία της κάλπης για σας είναι ήττα. Εσείς που εδώ στο Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πολλαπλασιάζετε τους χειρισμούς ε, για να αποφύγετε και να αποτρέψετε το Brexit. Και εσείς καμιά φορά ε, πάση θυσία θελήσατε να εγκριθεί ένα κείμενο που ήταν ε, απέναντι στη βούληση των λαών και στα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας και προφανώς απαράδεκτο για τη Βουλή των Κοινοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτών των ε, εκλογών ήταν διπλή νίκη για τον Μπόρις Τζόνσον. Πρώτον, δημοκρατική νίκη. Ε, έγινε σεβαστό το δημοψήφισμα, επέβαλε την απόφαση και την επιλογή του κυρίαρχου λαού και ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να βγει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι και πολιτική νίκη, γιατί ένωσε το λαό του, έδωσε στην πολιτική οικογένεια τη μεγαλύτερη εκλογική νίκη της τελευταίας 30 ετίας και ξεφορτώθηκε ε, θέματα όπως είναι αυτή η χαλάρωση στο μεταναστευτικό και ε, η παγκοσμιοποίηση κτλ. Ο Μπόρις Τζόνσον ε, πραγματικά είναι πάρα πολύ ε, στεναρός, ισχυρογνώμων και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού του. Θα έχουμε τώρα σχέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία που είναι μια μεγάλη χώρα σπουδαία, φίλη και σύμμαχος και δεν θα πρέπει να φοβούμαστε τον ανταγωνισμό γιατί ανταγωνισμό έχουμε και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των κρατών μας. One minute, Mr. Lundgren. Κύριος Λούγκρεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στην ουσία διάνθησε την ευρωπαϊκή συζήτηση σήμερα θα μας επιτρέψει να βάλουμε πίσω μας όλα αυτά τα θέματα. Όμως σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Τα προβλήματα των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή